Vielleicht war trochę z opóźnieniem. Można powiedzieć, że z kwadransem akademii. Γεια σας, ξεκινάμε με κάποια καθυστέρηση. Έχουμε ένα τέταρτο καθυστέρηση που είναι αποδεκτό ακόμα. Λοιπόν, όπως έλεγα, έχουμε μείνει λίγο πίσω. επιτρέψαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο να περάσει. Ίσως διότι και το θέμα μας είναι ακαδημαϊκής φύσεως. Είναι, έχουμε μορφή σεμιναρίο εργαστήριο με συζήτηση. Και είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύτιμο πολύτιμη συζήτηση. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Το δεύτερο τμήμα διαμόρφωσης πολιτικής, το οργάνωσε αυτό, είναι ένα εργαστήριο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στα πλαίσια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Η συνεδρίαση είναι και των θυρών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, ερευνήσει το θέμα των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ και το τμήμα πολιτικής πιστεύει ότι ένα εργαστήριο και κλεισμένο των θυρών θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες και στα μέλη εξίσου να προβούν σε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, ειλικρινή συζήτηση. Όλοι καλούνται να λάβουν το λόγο, όχι μόνο τα μέλη, και θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις όλων. Και υπάρχει και μια ομάδα έρευνας που, της οποίας ηγείται το κέντρο για τις ευρωπαϊκές ε, μελέτες και έχει ετοιμάσει το έργο αυτό για την Επιτροπή Γεωργίας. Λοιπόν, Εξετάζουμε την ιστορία της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει θέσει σε ισότιμη βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Η έρευνα εντασσόταν στις διευρυμένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να εξετάσουμε πώς αυτές οι διευρυμένες αρμοδιότητες έχουν επηρεάσει την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ποιες πτυχές. Ίσως σε αυτό το σημείο μπορώ να σχολιάσω εν συντομία ε, και τα όσα υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, τελειούν υποπίεση. Ε, μάλλον ήταν υποπίεση κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης και αυτό σημαίνει ότι είχαμε την εντύπωση ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να εγκρίνουμε κάποιες προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα βλέπουμε ότι ίσως τότε έπρεπε να είμαστε πιο αποφασιστικοί. πρέπει να είμαστε πιο αποφασισμένοι στις θέσεις μας τότε. Ε, αλλά είχαμε συνηθίσει, βλέπετε, ε, με τις ε, εξελίξεις του παρελθόντος και το κλίμα του παρελθόντος. Η χθεσινή ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο με οδήγησε να προβληματιστώ, να τα σκεφτώ όλα αυτά που σας ανέφερα. Να σας καλωσορίσω λοιπόν όλους σας και ακόμα και τα πρώην μέλη της ε, Επιτροπής Γεωργίας, τον κύριο George Lyon, Όλοι θυμόμαστε την περίφημη έκθεση Λάιον που ξεκίνησε την όλη συζήτηση και καθόρισε τις διάφορες ε, προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Και δεν ξέρω τι σημαίνει, τι συνέβη συγγνώμη μετά από αυτό, κύριε Λάιον. Νομίζω ότι κάπου ξεχάσαμε ε, να δούμε τα πράγματα από ευρύτερη οπτική γωνία. Φορούσαμε παροπίδες. Έχουμε και τον κύριο Καπούλα Σάντους εδώ μαζί μας. Έναν άλλον εισηγητή. Πάντα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε ε, εντελώς διαφορετικές απόψεις όμως ο κύριος Καπούλα Σάντους έκανε υπέροχη δουλειά κατάφερε να βρει μια ανθρώπινη ε, μορφή της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και να την περιγράψει στην έκθεσή του στους εμπειρογνώμονες Έχουμε και τον καθηγητή Γιώχαν Σουίνεν του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών Πολιτικής. Καλώς ορίσατε. Ο καθηγητής Σουίνεν θα μιλήσει πρώτος. Έχουμε και τον κύριο Ατίλα Κόβατς από το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας. Μετά θα διεξαχθεί η συζήτηση. Θα μας μιλήσει και ο κύριος Ντεκάστρο σαν πρώην πρόεδρος. Μετά θα ακούσουμε και τους πρώην εισηγητές της εποχής της μεταρρύθμισης, τον George Lyon, τον κύριο Καπουλοσάντους και τον κύριο Μισελ Νταντά. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Ντες θα μας μιλήσει. Νομίζω ότι είναι στο Βερολίνο ο κύριος Ντες σήμερα. Δεν είμαι σίγουρος. Αν ήδη έχει φύγει, πιθανότατα έχει φύγει ο κύριος Ντες. Μετά Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν είναι και ο κύριος Λαβία εδώ. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεν ήταν δυνατόν να είναι εδώ μαζί μας. Μετά από αυτή την, ε, μεγάλη εισαγωγή και ζητώ συγγνώμη που με μακριγόρησα αλλά όπως έλεγα είναι ακαδημαϊκό το θέμα μας και η συνεδρίασή μας Οπότε αισθάνομαι ότι έχω το δικαίωμα και εγώ να εκφράζω μεγαλόφωνα τις σκέψεις μου όπως έκανα στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό, αλλά ας μην χρονοτριβούμε άλλο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με αυτά που σας πρότεινα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Σουίνεν, ούτω ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες μας. Άλλη μόνησαν να καλωσορίσω κάποιον, σας παρακαλώ κάντε μου ένα ανέβημα, αλλά βασίζομαι και στη γραμματεία να με ειδοποιήσει ποιον θα καλωσορίσω. Ε, thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με παρουσιάσατε ως εμπειρογνώμονα στον τομέα αυτό, αλλά αισθάνομαι σήμερα το πρωί ότι είμαι λίγο εκτός τόπου, διότι νομίζω ότι οι εμπειρογνώμονες βρίσκονται εδώ στην αίθουσα και εγώ θα έπρεπε να ακούω αυτούς αντί να ακούνε αυτοί εμένα σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχω κάνει πολλή εργασία για την πολιτική και την οικονομία της κοινή αγροτικής πολιτικής και ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα έργα που έκανα, διότι μου ζήτησαν οι ίδιοι πολιτικοί να αξιολογήσω θέματα πολιτικής το θέμα το δεύτερο θέμα για το οποίο ήταν δύσκολο είναι επειδή το θέμα είναι δύσκολο, διότι μας ζητήθηκε ε, να αξιολογήσουμε την μοναδική εμπειρία. Μοναδική εμπειρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκρισης, δεν υπήρχε ε, ε, περίοδος κατά την οποία να είχε συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα τέτοιο θέμα και αυτό που ήταν επίσης πρόκληση εδώ δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα πρότυπα, τα σημεία αναφορά, τα benchmarks για να συγκρίνουμε ε, την ε, απόδοση, τα αποτελέσματα, ποιο ήταν το επίπεδο των άμεσων πληρωμών που είχαν αποφασιστεί, αν ήταν καλές, αν ήταν κακές ε, ήταν λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση. Επίσης το timing, ο χρόνος, ο χρονισμός. Είχαμε τέσσερις μήνες για ολόκληρη την μελέτη, αλλά βεβαίως η έρευνα ε, συνήθως χρειάζεται συλλογή, διεκπαιρέωση, ε, επεξεργασία δεδομένων, ένα πλαίσιο θεωρητικό. Είναι σαν να παράγει κανείς κρασί το κρασί γίνεται καλύτερο όταν περνάει ο χρόνος, όταν ε, γυρνάει το κρασί. Ε, ήταν, έπρεπε λοιπόν σαν την μπύρα να, να κάνουμε αυτή τη δουλειά, η οποία η μπύρα είναι ένα φρέσκο προϊόν. Πάντως αυτό που θα έχετε σήμερα είναι κάτι για το οποίο όλοι θα συμφωνήσετε είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί με περαιτέρω εργασία, με ορίμανση αν θέλετε, με συζήτηση και νομίζω ότι αυτό ισχύει κυρίως στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης σχετικά με τα βασικά διδάγματα και συστάσεις που μπορούμε να εξαγάγουμε βάσει της έκθεσης. Νομίζω ότι είναι μάλλον ιδέες για συζήτηση και όχι τελικές συστάσεις. Για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις έχω ε, μια, ένα συνδυασμό των ε, διαφόρων ερευνών, νέων ερευνητών που κάθονται δίπλα μου, ε, με επίσης μια ομάδα παρακολούθησης μεγαλύτερων για να δείξουμε την δυναμική και για να έχουμε ένα προϊόν νέο αλλά καλό. Επίσης εδώ έχουμε ε, το μείγμα και θα ήθελα να κάνω το πρώτο μέρος παρουσίασης και το τέλος ε, της παρουσίασης, ε, ενώ οι αυτοί που κάθονται δίπλα μου θα ασχοληθούν με τα δύσκολα θέματα. Θα κάνω λοιπόν ανάλυση των τροπολογιών και ο Άλαν Μάθιους που όλοι γνωρίζετε έχει ασχοληθεί με μια μελέτη παραδείγματος και θα κάνει και μια σύντομη παρουσίαση σε βίντεο. Έχουμε το, το αποτέλεσμα πολύ ε, μακρύτερο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Υπάρχουν τέσσερις εκθέσεις ε, βασικές που είναι διαθέσιμες και θα εξηγήσω ε, τι είναι αυτές οι βασικές εκθέσεις, οι background reports και στην παρουσίασή μου θα τονίσω μερικές από τις διαπιστώσεις και θα, στο, στη βασική έκθεση θα έχουμε τις λεπτομέρειες. Πρωτού αρχίσω θα ήθελα να ευχαριστήσω μερικά άτομα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα διότι με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα με την ομάδα με πολλή ενθάρρυνση και επίσης είχαμε και επικρίσεις για τα όσα κάναμε και Είχαμε την τεχνική βοήθεια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς από εσά που αφιέρασαν χρόνο και γνώσεις για συνεντεύξεις και επεξεργασία και ευχαριστώ το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ε, που εξέτασε τις δύο προκαταρκτικές εκδοχές της έκθεσης και που έκανε κριτικές και χωρίς την βοήθεια του προσωπικού δεν θα ήταν εφικτό αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ σύντομα σε σχέση με την παρουσίαση έχουμε πέντε τμήματα αν θέλετε θα ασχοληθώ με τους στόχους και την μεθοδολογία, θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα της ανάλυσης τροπολογιών και μερικά πιο γενικά αποτελέσματα. Ο Άλαν Μάθιους θα σας μιλήσει για μια, ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα τρία βασικά ερωτήματα ήταν πώς η συναπόφαση επηρέασε την μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ του 2013, εάν οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άσκησαν την μέγιστη επιρροή και πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει την μελέτη. Η προσέγγιση μας εστιάστηκε στην εσωτερική δυναμική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην διαθεσμική δυναμική ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά ε, όργανα, πώς οι εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν όλα αυτά τα πράγματα και μετά ποιοι παράγοντες και άλλα στοιχεία έχουν ή περιορίσει ή ενθαρρύνει την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον και επίσης η μεγαλύτερη ε, πρόκληση ηταν ενδιαφερον και επισης αμεγαλύτερη ότι η ΠΑΚ της 2013 συζητήθηκε όταν γινόντουσαν πολλά πράγματα στον κόσμο. Είχαμε την μεγαλύτερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 30, είχαμε αλλαγή της οπτικής ε, της τροφικής ασφάλειας λόγω των τιμών ε, των τροφίμων, είχαμε ε, πολλά νέα κράτη-μέλη τα οποία προσχώρησαν ε, στην κοινή αγροτική πολιτική που δεν ήταν πριν μέλη και είχαμε τις αποφάσεις ε, για τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα σύνολο παραγόντων πάρα πολύ περίπλοκο μέσα στο οποίο πλαίσιο έπρεπε να υπάρξει αυτή η συναπόφαση. σχέση με την βιβλιογραφία δεν είχαμε τόση πολλή βιβλιογραφία διότι οι μελέτες που προϋπήρχαν δεν μπορούσαν ήταν εξάντ και είχαν προβλέψει τι θα συνέβαινε, αλλά καμιά από αυτές τις μελέτες δεν είχε αναλύσει ε, τι είχε γίνει. Είναι η πρώτη μελέτη που προσπάθησε να το πράξει. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε ήταν ρεαλιστική για πολλούς λόγους, επίσης λόγω ε, του χρονικής περίοδου και της πίεσης. Είχαμε συνεντεύξεις ατόμων, θα εξηγήσω περισσότερα γι' αυτό, ανάλυση τροπολογιών που θα εξηγηθεί και μετά τέσσερις μελέτες που έγιναν για ε, βασικά ε, θέματα. Η ε, δυναμική της Κομάγκρη, το πρασίνισμα, το οικολογικό, το ρόλο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και το θέμα της ρύθμισης της αγοράς. Και όλες αυτές οι μελέτες είναι ξεχωριστή μελέτη και είναι διαθέσιμη. Είχαμε, ε, πήραμε συνεντεύξεις από 34 ε, βασικούς πρωταγωνιστές, άτομα που είχαν εμπλακεί στη συζήτηση και στις μεταρρυθμίσεις. Μεταξύ 30 λεπτών και 2 ώρες ε, οι συνεντεύξεις πλήρης ανωνυμία όλων των ατόμων που ερωτήθηκαν. Το ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε και ε, στείλαμε στα άτομα που ερωτήσαμε μια, ένα αντίγραφο, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι ήταν σωστές οι απαντήσεις. Στην σελίδα 25 έχετε τις συνεντεύξη στα άτομα από τα οποία πήραμε συνέντευξη, από πού προέρχονται, επειδή βεβαίως ε, υπάρχει ανωνυμία, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τα στοιχεία τους, ε, πόσοι από ένα θεσμικό όργανο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών ε, και επίσης εξωτερικοί παρατηρητές. Όσον αφορά την ανάλυση τροπολογιών, ε, θελήσαμε να, μετρήσουμε, να σταθμίσουμε την νομοθετική επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, να δούμε και βεβαίως ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα, αν, είχαν, ενσωματώθηκαν οι τροπολογίες ε, και έχουμε λοιπόν πολλά, πάρα πολλά στοιχεία, είδαμε τον βαθμό επιτυχίας και κάναμε διάφορες συγκρίσεις. Θα δώσω τώρα τον λόγο για να σας δώσει μερικά αποτελέσματα ο Άλαν. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε όλοι. Να αναφερθώ εν συντομία στα βασικά αποτελέσματα των τροπηγιών, των αναλύσεων κλπ. Και τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε οδηγίες για την κοινή πολιτική, λέξαμε όλες τις τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης τροπολογίες στις γνωμοδοτικές επιτροπές και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην Ολομέλεια. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρία στάδια στην ανάλυση αυτή. Ε, είδαμε κατά πόσο εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων, αν εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο Ολομέλειας και το τρίτο σημείο κατά πόσο οι τροπολογίες αυτές μπήκαν στο τελικό κείμενο της νομοθεσίας. Η ανάλυση μας επίσης έχει και μία σύγκριση σε επίπεδο της διαδικασίας συναπόφασης. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τον αριθμό των τροπολογιών που κατατέθηκαν για τους τέσσερις κανονισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής το κύριο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από αυτή τη ε, διαφάνεια είναι ο μεγάλος αριθμός <clears throat> των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Αυτό σημαίνει ότι ίσως ότι οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι αυτοί θα πρέπει να επηρεάσουν περισσότερο τις προτάσεις της Κομισιόν. Δεύτερον, την ε, με τη διαδικασία διαβούλευσης οι περισσότερες τοπολογίες είχαν να κάνουν με, την, ε, με τον κανονισμό άμεσων πληρωμών ενώ μετά την ε, μεταρρύθμιση με την συναπόφαση είναι κάπως πιο ισορροπημένη η κατανομή των τροπολογιών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την κατανομή των τροπολογιών όχι μονάχα επί τη βαστού κανονισμού αλλά και για το είδος τροπολογιών. Η τροπολογίες στο σχέδιο έκθεση είναι αυτές που έχουν ενσωματωθεί στην έκθεση του εισηγητή, οι ανοιχτές τροπολογίες είναι αυτές που έχουν κατεθεί από άλλους βουλευτές. Οι τροπολογίε των γνωμοδοτικών επιτροπών είναι αυτέ που βλέπετε εδώ. Οι συμβαστικέ τροπολογίε επίση ε, καταγράφονται χωριστά. Υπήρχαν κάποιε τροπολογίε προφορικού χαρακτήρα και κάποιε τροπολογίε στην Ολομέλεια. Βλέπετε ότι περισσότερες περισσότερε τροπολογίε είναι οι ανοιχτέ τροπολογίε. Και πολύ λίγες από αυτές ήταν πραγματικά ουσιαστικές και μπήκανε στις συμβαστικές τροπολογίες. Εδώ βλέπουμε μια γενική επισκόψη του ποσοστού επιτυχίας στα τρία αυτά στάδια τα οποία ανέφερα. Πιο σημαντικά στοιχεία εδώ είναι το ότι 10 περίπου τα 100 των τροπολογιών εγκρίθηκαν τελικά, μπήκαν στον τελικό κανονισμό και στη διαδικασία διαβούλευση στο παρελθόν και με την συναπόφαση τώρα. Κάπως λιγότερο στην προηγούμενη διαδικασία, κάπως περισσότερο με την συναπόφαση. Αν θυμόστε την προηγούμενη διαφάνεια, 10% σημαίνει περίπου 140 τροπολογίες οι οποίες ενσωματώθηκαν στον κανονισμό βάση της διαβούλευσης, ενώ το 10% στην περίοδο της συναπόφασης σημαίνει περίπου 900 τροπολογίες. Και ξαναδίνω στον κύριο Σουίνεν τον λόγο. Τα υπόλοιπα στοιχεία της έκθεσης. Εδώ είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι, το κομμάτι των πορισμάτων της έκθεσης. το κεφάλαιο 4. Τι έγινε στην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συναπόφαση. Το πέμπτο τι έγινε μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6. ποια ήταν η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτά τα τέσσερα σημαντικά θέματα που ανέφερα και μετά περνάμε στο πώς επηρεάστηκε Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο το θέμα στο κεφάλαιο 4. Αυτά που κοιτάξαμε λοιπόν για την εσωτερική δυναμική είναι ποια είναι η σύνθεση της Επιτροπής Γεωργίας, ποιος είναι ο ρόλος των εισηγητών, ποιες είναι οι εσωτερικές ε, ισορροπίες και η δυναμική ποια είναι η πόρη της Επιτροπής Γεωργίας, ποια είναι η φύση της Επιτροπής Γεωργίας για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος είναι ο ρόλος των γνωμοδοτικών επιτροπών και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών στην Επιτροπή Γεωργίας και στην Ολομέλεια. Θα σας δώσω λοιπόν μερικά πολύ κέρια αποτελέσματα εν συντομή και σας ζητώ συγγνώμη γιατί πολλά από τα συμπεράσματά μας πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφοροποιημένο τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε ιδιαίτερα σαφή αποτελέσματα. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή Γεωργίας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην λήψη απόφαση σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικά. Ένα από τα πορίσματά μας είναι ότι στην απόφαση δεν άλλαξε τη φύση της σύνθεσης Επιτροπής Γεωργίας. Αυτό περιμένουν κάποιοι εμπειρογνώμονες εκ των προτέρων, γιατί θεώρησαν ότι με τη μεγαλύτερη ε, δυνατότητα συναπόφασης θα ήταν και άτομα τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς που θα θέλουν να μπουν στην Επιτροπή Γεωργίας και αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε. Δεύτερον, προφανώς οι συγητές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία υπήρξε κάποια συζήτηση, δεν συμφωνήσαν όλοι για το κατά πόσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο η κατανομή των εκθέσεων. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος εισηγητής για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη συζήτηση με τους εξωτερικούς φορείς και συντονισμό. Άλλοι λέγαν τέσσερις εισηγητές. Γενικά, πρέπει να πω ότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά μεγάλη εκτίμηση για το έργο των εισηγητών. Επίσης μπόρεσε να καταλήξει συμφωνίες η Επιτροπή Γεωργίας. Αυτό δείχνει την ικανότητα να ξεπεραστούν οι πολιτικές διαιρέσεις μέσα και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αλλά βέβαια στη διαδικασία συναπόφασης ήταν πιο έντονες οι διαφοροποίησεις. Παρά το γεγονός ότι κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση. Ματήρα ανέφερε για τον, ε, προηγουμένως για τον ρόλο των γνωμοδοτικών επιτροπών. Και τώρα φυσικά με την τεχνολογική καινοτομία είναι πολύ πιο εύκολο να καταθέσει κανείς τροπολογίες από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα οι άλλοι κοινοβουλευτικοί φορείς και η επιρροή τους. Εδώ υπήρξε συνένεση ότι οι γνωμοδοτικές επιτροπές είχαν περιορισμένη επιρροή λιγότερο από ό,τι μπορεί να θεωρούσαν καταρχήν οι εξωτερικοί παρατηρητές. Προφανώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν η πιο ενεργή από τις επιτροπές, αλλά ήταν αρκετά έντονη η σχέση της Επιτροπής Γεωργίας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τελικά ήταν περιορισμένος ο αντίκτυπος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το θέμα τώρα του σε ποιο βαθμό πόσο μεγάλη είναι η επιρροή στις ε, Επιτροπές Γεωργίας σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε λιγότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, αυτή είναι η γενική εικόνα, αλλά είναι δύσκολο να το πει κανείς γενικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που η Επιτροπή Γεωργίας προχώρησε περισσότερο από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και φυσικά το πιο δύσκολο και συγκινησιακό θέμα ήταν το θέμα του πρασινίσματος. Επίσης, οι διαφορές μεταξύ της απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και της Ολομέλειας ήταν γενικά μικρές, κάποιες φορές διαφορετικοί. Και στην Ολομέλεια πολλές φορές η εθνική προέλευση ήταν πιο σημαντική από την κομματική τοποθέτηση. Ένα σημαντικό θέμα και για το μέλλον είναι η αυξανόμενη ευθύνη της ε, συναπόφασης δεν οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των πόρων που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ υπήρξε αυτή η σχέση πολιτικής επιρροής και τεχνικών δυνατοτήτων για την Επιτροπή Γεωργίας. Περιμέναμε ότι περισσότεροι πόροι, κυρίως τεχνολογικές δυνατότητες, θα έδιναν μεγαλύτερη δυνατότητα στην ε, διαπραγματευτική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ρωτήσαμε πολλούς ποια ήταν η άποψή τους για το μέλλον και δεν υπάρχει ευρεία συνένεση. Είπαν οι περισσότεροι, καλό θα ήταν να είχαμε κάπως περισσότερους πόρους αλλά δεν θεωρούν ότι πρέπει να φτάσει στο επίπεδο της Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζεται ως ε, ένας φορέας ο οποίος μπορεί να δώσει εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον. Κεφάλαιο 5. γονικοί διάλογοι. Δώσαμε διάφορα σενάρια στους ερωτώμενους για να μας πούν ποια ήταν η άποψή τους ποιο σενάριο επικρατεί για τη διαδικασία συναπόφασης. Γενικά όλοι ακολούθησαν τους Greer και Hind το συμβατικό αυτό σενάριο που λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κέρδισε εξουσία σε βάρος των άλλων θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι εδώ το αναγνωρίζουν όλοι. Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικός νομοθέτης και έχει γίνει ένα ενεργό κοινοβούλιο για την κοινή αγροτική πολιτική. Επομένως, δεν είναι ένα δεύτερο κοινοβούλιο που απλώς επικυρώνει αυτά τα οποία λέει το Συμβούλιο, αλλά ήταν πάρα πολύ ενεργός και ε, με επιρροή παίκτη σε αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό επίση ότι υπάρχει μια νέα κουλτούρα εργασίας που πολλέ φορέ ήταν επιτυχημένη αλλά όχι πάντα. Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και η αναγνώριση του ρόλου των οργάνων αυτών. Οι άτυπες επαφές είναι κέρδιες και αυτό το αναγνώρισαν όλοι μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το λάβουμε υπόψη και για το μέλλον υπάρχουν πιο έντονες επαφές μεταξύ μη θεσμικών εμπλεκομένων. Αυτό είναι θετικό από τη μία πλευρά. Γιατί μπορεί η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει και οι εμπλεκόμενοι στα θέματα αυτά, αλλά συγχρόνως υπάρχει το θέμα του κατά πόσο με περιορισμένους εσωτερικούς πόρους η αλληλεπίδραση αυτή με τους, με τους εξωτερικούς φορείς κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ευάλωτο ή την Επιτροπή Γεωργίας πιο ευάλωτο στην επιρροή αυτών των εξωτερικών φορέων. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως είναι και η επιτυχία της Ιρλανδικής Προεδρίας και αυτό δεν είναι μια αυτόνομη επιτυχία, είναι και ένα <coughs> δείγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσει θετικά η συναπόφαση. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι, ότι η ελληνική Προεδρία επένδυσε πολύ σε μια προσωπική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό δείξε σε μια σημαντική επιρροή του τελικού αποτελέσματος. Επίσης υπάρχει και το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εκεί μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στο μέλλον με νέες θεσμικέ διευθετήσεις ή προσαρμογές, ούτως ώστε όλα αυτά να προβλέπονται και να προλαμβάνονται. Όσον αφορά την επιρροή, προφανώς όπως ανέφερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει νέες εξουσίες και έχει μεγαλύτερη επιρροή στη συναπόφαση από ό,τι πριν περιορισμένους τεχνικούς πόρους που ίσως περιορίσουν όμως την επιρροή. Δεν ξέρουμε πώς επηρέασε εξουσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να είναι διευκολυντής και να δίνει τεχνογνωσία και έτσι μπορούσε να, να επηρεάσει τις εξελίξεις αλλά έχει λιγότερη επιρροή τώρα κυρίως εκεί που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν συμμαχήσει, έχουν συνασπισμό για κάποιες θέσεις και στην ανάλυση των τροπολογιών το βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο συνεργάζεται καλύτερα με το Συμβουλίο και εκεί που ενώνουν τις δυνάμεις τους ήταν πάρα πολύ επιτυχής. Ο Ατήλα ίσως θα μας δείξει κάποιες, ε, ε, κάποια αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της αναλύσεως των τροπολογιών. Βλέπουμε λοιπόν τα ποσοστά επιτυχιών των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ολομέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι τους τελικούς κανονισμούς στους τριγωνικούς διαλόγους. Στη διαδικασία διαβούλευσης περίπου 30% σχεδόν διπλασιάστηκε στην συναπόφαση εν γέννη. Ε, it's to note. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποια επιρροή και στα πλαίσια της διαβούλευσης μπορούμε να συζητήσουμε για ποιους λόγους δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες, υπάρχει κάποια επιρροή. Στη συναπόφαση αυξήθηκε. Αν δούμε τα στοιχεία, βλέπουμε ότι όσον αφορά την αλλαγή των τροπολογιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ισχυρότερο. Στα πλαίσια του κανονισμού EAFRD και χαμηλότερο ποσοστό είναι στο του κανονισμού εν γέννη. Οι περισσότερες επιτυχίες είναι στο EAFRD δεύτερον οι άμεσες πληρωμές και ο κανονισμοί CSMO και στη τρίτη θέση είναι οριζόντιος κανονισμός. Δεν θέλω να τερμινεύσω αυτά σαν την, ότι αφορούν το βάρος ή την εξουσία ή τη δύναμη των εισηγητών. Αν ενδιαφέρον ε, να δούμε πόσο μπορούσαν να επηρεάσουν και οι εισηγητές εξελίξεις. Δεύτερη, επόμενη διαφάνεια βλέπετε στοιχεία ανάλογα με το είδος των τροπολογιών και εδώ μπορούμε να συναγάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το πρώτο που τονίζω είναι το εξής. Οι περισσότερες επιτυχίες ήταν στις συμβαστικές τροπολογίες. Από τη στιγμή που ενταχθεί σε συμβαστική τροπολογία, μια τροπολογία, η πιθανότητα προσέγγιση συμβιβαστικής και των συγχωνευμένων αρχικών ε, τροπολογιών είναι αυξημένε. Άλλο συμπέρασμα. Οι επιτροπές που γνωμοδοτούν έχουν περιορισμένη επιρροή στο αποτέλεσμα πολιτικής. Τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχιών είναι στις επιτροπές που γνωμοδοτούν. Ε, να σημειώσουμε τώρα ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν η πλέον δραστήρια στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει υποβάλει περισσότερες τροπολογίες ε, νομοθετικού περιεχομένου, αλλά όσον αφορά τις επιτυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ήταν η πλέον επιτυχής. Όμως οι τροπολογίες της δεν ήταν απαραίτητα σχετιζόμενες με διαμόρφωση πολιτικής, αλλά με ε, εμπορικά θέματα, σχέση με τίτες χώρες κλπ. Η τροπολογία στην Ολομέλεια για όλες τις τροπολογίες τα ποσοστά επιτυχιών έχουν διπλασιαστεί και σε κάποιες περιπτώσεις ε, πενταπλασιαστεί, εξαπλασιαστεί τα ποσοστά επιτυχίας. Οι ανοιχτές τροπολογίες Λοιπόν, τα σχέδια τροπολογιών και λοιπά σχετίζονται και με το βάρος και την επιρροή των ε, εισηγητών. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο καθηγητή. Το κεφάλαιο 6 έχει τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα για συγκεκριμένα θέματα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ανώτατα όρια, το πρασίνισμα, ε, επιρροή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και τις διάφορες προτάσεις. Θα δώσω το λόγο στον Άλαν Μάθιους που έστειλε βιντεοδήλωση όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη τη Επιτροπή, καλημέρα. Το όνομά μου είναι Άλαν Μάθιου και είμαι καθηγητή ε, που διδάσκει Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική στο Trinity ε, College στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία. Αξιολογώντα τον αντίκτυπο τη συναπόφαση στην πρόσφατη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ, ένα σημαντικό στοιχείο ήταν οι παράλληλε διαπραγματεύσει όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Σε μία από τις μελέτες περιπτώσεων που ετοιμάστηκε σαν ένα πρόγραμμα του προγράμματο ενετόπισα τρει διασυνδέσει μεταξύ των διαπραγματεύσεων που είχαν ε, επηρέασαν κάπω το αποτέλεσμα. Η πρώτη σχέση ήταν όσον αφορά τη φάση καθορισμού του προγράμματο μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Η Γενική Διεύθυνση Άγκρη έκανε μια πρόταση που αιτιολογούταν από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν νέε προκλήσει που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Γεωργία στην Ήπεθρο. Επίσης και η ανάγκη να δημιουργηθεί μια προσέγγιση που θα βοηθήσει να υπερασπίσει κανείς και να βυθιστοποιήσει τον προπολογισμό της ΚΑΠ σε διαπραγματεύσεις εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που θα πρότεινε. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρηθεί ο προπολογισμό τη ΚΑΠ στα επίπεδα του 2013 σε ονομαστικού όρου σαφώ επηρεαζόταν από τι προσδοκίε ότι η νέα ΚΑΠ θα εστιαζόταν πολύ περισσότερο σε περιβαλλοντικού στόχου από ό,τι κατά το παρελθόν. Δεύτερη διασύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω του προγραμματισμού των δύο ε, διαπραγματεύσεων. Από την αρχή το Κοινοβούλιο είπε ότι δεν θα ήταν έτοιμο να θωμοτήσει για μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ μέχρι ότου είχαμε γνωστά στοιχεία για τον προπολογισμό. Η καθυστέρηση από πλευρά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για οριστικά στοιχεία για το πολιτέ πλαίσιο μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 είχε δύο συνέπειε. Πρώτη συνέπεια, συμπίεσε τον διαθέσιμο χρόνο για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει για την ΚΑΠ, δοθήσει στι προτιμήσει όλων των μερών τη μια συμφωνία θα έπρεπε να επιτευχθεί πριν το τέλο τη Ιρλανδική Προεδρία τον Ιούνιο του 2013. Όμω Όμως δεν υπάρχει σαφές στοιχείο ότι η μακρύτερη περίοδο για τους τριγωνικούς διαλόγους θα άλλαζε το αποτέλεσμα η θα οδηγούσε σε διαφορετική συμφωνία. Και, ότι, και πιο σημαντικό η αιμονή του Κοινοβουλίου ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσει σοβαρέ διαπραγματεύσει για την ΚΑΠ μέχρι ότου ήταν γνωστά τα ποσά του προπολογισμού ευνόησε εκείνους που ήθελαν να διατηρηθεί ε, το status quo όσον αφορά τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση, ενώ έφερε σε δυσχερή θέση εκείνους που θέλανε πιο ριζοσπαστικέ αλλαγέ όσον αφορά τον προσανατολισμό της ΚΑΠ. Από τη στιγμή που εθετήθηκε το, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το γενικό μέγεθο και τα Νότατα όρια έγιναν αποδεκτά από το Κοινοβούλιο στι αρχέ του 2013, η απειλή ενό υπολογισμού που θα περιεκόπτετο και θα αποδυναμωνόταν το υπρασίνισμα δεν έπαιξε κανένα ρόλο στον καθορισμό του αποτελέσματο. Έτσι, ομάδε γεωργών και διάφορα κράτη-μέλη και ευρωβουλευτέ μπόρεσαν να αποδυναμώσουν τη φιλοδοξία των προτάσεων για το πρασίνισμα χωρί να ανησυχούν να το οδηγούσε σε μία μείωση του προπολογισμού για την ΚΑΠ ε, που έτσι το ερμήνευε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν η τρίτη, τρίτη σχέση μεταξύ του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου και των υπερκοθέσεων για το ΚΑΠ που έθεσε το θέμα ε, τη συναπόφαση. Αυτό ήταν η συμπερίληψη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το πολιτικό δημοσικό πλαίσιο θεμάτων που τελικά θα έπρεπε να ενσωματωθούν στους νέους κανονισμούς περί ΚΑΠ που θα αποφασιζόταν μέσω συναποφάσεως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί επουσιαστικών θεμάτων πολιτική. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αμφισβητεί κανεί. Η δυσκολία όμω προέκυψε διότι τα θέματα που συμπεριέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του ε, απέκτησαν προνομιακή θέση από πλευρά των διαπραγματευτών του Συμβουλίου στι τριγωνικέ συνομιλίε. Το Κοινοβούλιο κέρδισε κάποιε παραχωρήσει στην τελική διευθέτηση, όμω ο ρόλο του σαν συνομοθέτη σε αυτά τα θέματα μειώθηκε. Αυτό είναι σίγουρο. Το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να περάσει κάποιε τροπολογίε και να αλλάξει θέσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σημαντικό σημείο να ληφθεί υπόψη μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Παρ' όλα αυτά, Θεωρώ ότι η εξουσία του Κοινοβουλίου να επηρεάσει την νομοθεσία μέσω συναπόφαση αναπόφευτα θα περικοπεί σε περιπτώσει όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θετηθεί ομόφωνα. Ιδιαίτερα, κάνω διάκριση μεταξύ των νομοθετικών αποφάσεων για την ΚΑΜ που άμεσα επηρεάζουν τι ροέ από τον προπολογισμό των Ευρωπαϊκών προ τα κάτι μελη παραδείγματο χάρη η εξωτερική σύγκληση ή η διανομή των πληρωμών του πυλώνα 2 και άλλα νομοθετικά θέματα. Ε, λέω ότι το Κοινοβούλιο πάντα θα θεωρεί ότι είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξουν οι ομόφωνες ε, ε αποφάσεις των αρχαιών κρατών κυβερνήσεων όσον αφορά την άμεση διάθεση των πόρων. Και το συμπέρασμά μου είναι ότι αν το Κοινοβούλιο θέλει να επηρεάσει αυτή την κατανομή των πόρων, τότε θα πρέπει να ασκήσει αυτή την επιρροή πριν ε, καταλήξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συμπεράσματα. Από την άλλη πλευρά, όλα άλλα τα θέματα που σχετίζονται με την ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πλήρω ανεκτά στι τριγωνικέ διαπραγματεύσει ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα. Σα ευχαριστώ. Okay, let me then τότε θα ήθελα απλώς να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι και μετά θα πρέπει να σας δώσουμε σας το λόγο για την συζήτηση. Έχουμε λοιπόν αυτές, αυτές τα συγκεκριμένα παραδείγματα για ειδικά θέματα και είναι μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο προφανή όσον αφορά ε, το ημερολόγιο, όσον αφορά τον χρόνο για τις ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, θεωρεί το, το, αρχικό ημερολόγιο ως μη ρεαλιστικό για την, την διαδικασία διαμόρφωσης της ΚΑΠ. Επίσης το θέμα των προσδιορισμού ανωτάτου ορίου και το πρασίνισμα η αντίληψη του ρόλου που παίζει η συναπόφαση ε, πως οι άνθρωποι αισθανόντουσαν ότι το πρασίνισμα αυτό το οικολογικό ήταν επιτυχημένο ή δεν ήταν επιτυχημένο. Υπάρχουν διχογνωμίες ως προς το γεγονός αυτό. Μετά όσον αφορά το άρθρο 43.3 ε, νομίζω είναι παρόμοιο το σημείο με το σημείο που ανέφερε ο Άλαν σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η κατάσταση του Κοινοβουλίου ε, για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά την σφαιρική, την γενική αξιολόγηση, είχαμε το γεγονός ότι καταλήξαμε σε συμπέρασμα με, το, ε, με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι η συναπόφαση λειτουργεί καλά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Επίσης είχαμε έναν καλό βαθμό. Ε, ζητήσαμε να βαθμολογήσει κανείς, ε, να βαθμολογήσουν από 1 ως 7 ε, τη συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι 69%, 4,8 στα 7 βαθμό, είναι διάκριση στο Πανεπιστήμιό μου. Και αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον στην ανάλυση μας και στην έκθεση είναι ότι το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο είχε υψηλό βαθμό, αλλά από το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν επίσης. Ε, εκεί η κατάσταση ήταν αρκετά καλή. Είναι καλή εκτίμηση της εργασίας που έγινε όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα. Πολύ ανέφερα ότι υπήρχε αύξηση της λογοδοσίας, της διαφάνειας της διαδικασίας μεταρρύθμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης θα είναι εύκολο να αξιολογηθούν τα στοιχεία της επιτυχίας της συναπόφασης είναι πέντε κατά τη γνώμη μου, που εξήχθησαν από την μελέτη ευξημένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ένα σχετικά καλό περιβάλλον εργασίας ε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με άλλες και σε άλλα θεσμικά όργανα. Υπάρχει βεβαίως παντού ε, περιθώριο βελτίωσης, όλο το ανέφεραν σε σχέση με άλλες διαδικασίες. Βεβαίως εδώ έχουμε μια θετική εμπειρία υπάρχει μια κουλτούρα συμβιβασμού που είναι πολύ πιο ισχυρή. Επίσης αναφέρθηκαν πολλές φορές οι επιτυχημένες συναντήσεις σκιωδών ε, εισηγητών και ε, οι τριμερείς επίσης. Άλλα διδάγματα ή άλλα σημεία για το μέλλον είναι ότι τα άτομα παίζουν σημαντικό ρόλο, ε, οι συγητές, οι οι συγητές, οι ομάδες στήριξης, ε, το Προεδρείο κλπ. Η προετοιμασία και η επικοινωνία θεωρήθηκαν κάτι το σημαντικό και αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον, να αρχίζουμε αρκετά νωρίς και να μην περιμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής όσο το δυνατόν νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Η εκμάθηση με την πράξη, στην πράξη, με την πρακτική βεβαίως ήταν η πρώτη φορά και εσείς αντλήσατε τα δικά σας διδάγματα και ένα άλλο σημείο είναι ότι το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ παρά μόνο όταν τελειώσει πραγματικά υπάρχουν τα, οι συμβιβασμοί, υπάρχουν οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Έχω άλλη μια διαφάνεια νομίζω. Μερικά άλλα θέματα εδώ. Εγώ αναφέρα ήδη όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρονται στη διαφάνεια. Το θέμα της προσαρμογής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον νέο νομοθετικό ρόλο του είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί για το μέλλον. Και πάλι για να κλείσω, ήταν μια μελέτη πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη και ήταν στο μέσο της δράσης και έπρεπε να δούμε τα πράγματα απ' έξω ε, και το, η μελέτη αυτή έχει υλικό ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για το μέλλον. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρουμε σε πέρα σε αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Είναι πολύ δύσκολο να ερευνήσει κανεί. τι θέλει να κάνει το Συμβούλιο, τι θέλουν να κάνουν τα μέλη του Κοινοβουλίου, τι κάνει η Κομισιόν. Ο υπουργό Γεωργίας τη Ιρλανδίας είχε εμπειρία ως ε, ευρωβουλευτής. Και αυτό βοήθησε πολύ τη σχέση της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια πρέπει να πω ότι μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε μονάχα μισή ώρα μπροστά μας. Ο κύριος Κάστρο, Δεκάστρο, Λάιον, Καπόλα Σάντους, τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον καθηγητή Σόναν, τον κύριο Κόβακ, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά του σήμερα. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που διαβάσαμε στην ανάλυση για τις εργασίες μας για την μεταρρύθμιση. Καινοτόμως η προσέγγιση. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Θα να κάνω και εγώ σήμερα τον καθηγητή διότι είμαστε σε κεκλεισμένο το συνεδρίαση. Πάνω απ' όλα ένα στοιχείο. Είναι η πρώτη μεταρρύθμιση που πραγματοποίησαμε χωρίς έναν οικονομικό πλαίσιο. Αξιοσημείωτο. Θυμάμαι πολύ καλά το, την ε, αναθεώρηση της ατζέντα του 2012 του Φρανς Φίσλερ που επέβαλε μια απόφαση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τους δημοσιονομικούς πόρους πριν την αρχή των υπραγματεύσεων δεν θεωρώ ότι μπορεί να διαπραγματευτεί με μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ, λέω για το 1999, χωρίς ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήταν η πρώτη περίπτωση που ξεκινήσαμε στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουμε βεβαιότητα από αυτού. Το είπατε. Αυτό επηρέασε τα πράγματα πάρα πολύ. Όπως έλεγε η καθηγητή σου είναι, ουσιαστικά υπήρξε αύξηση της νομιμότητας της πολιτικής που προερχόταν από το πρασίνισμα, το greening. Το greening όπως είπατε είχε συναδέλφους που το υποστήριζαν περισσότερο, άλλους λιγότερο. Δεν ήταν θέμα τι πρασίνισμα θέλαμε. Ήταν θέμα τι πρασίνισμα θέλαμε, όχι αν θα υπάρξει πρασίνισμα. Και θέλαμε να δούμε αν αυτό το πρασίνισμα που είχαμε εισάγει, αν θα οδηγούσε στα περιβαλλοντικά ωφέλη που θα δικαιολογούσαν τις θυσίες θυσίες γραφειοκρατικές για τα κράτη-μέλη, θυσίες όσον αφορά το κόστος που συνεπέφερε. Δεύτερο στοιχείο που ίσως δεν υπογραμμίστηκε αρκετά ήταν η δυσκολία. Οι συνάδελφοι, ο Λούις Καπούλας, Μαγκίνες, Νταντέν και λοιπά και άλλοι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε αυτό το τομέα που είναι άκρος ενδιαφέρον στην προσπάθεια μεταρρύθμισης που έγινε, ο Τζορτζ Λάιν επίσης, το γνωρίζουν ότι ποτέ δεν καταφέραμε να μπούμε στο σωστό κλίμα με τον Επίτροπο. Δεν ξέρω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά κουραστήκαμε πολύ. Εγώ μπορέσα να συνεργαστώ με διάφορους επιτρόπους στη ζωή μου. Ο κύριος Τσόλος ήταν επίτροπος με τον οποίο στις τόσες συναντήσεις που είχαμε ποτέ δεν καταφέραμε να πετύχουμε, να έχουμε άμεση επαφή η έκθεση του George Lyon και του Albert Dess που ακολούθησαν όσον αφορά την πρόταση μεταρρύθμισης ποτέ δεν χωνεύτηκαν τους ΥΠΗΝ εντός ε, του γραφείου και του Επιτρόπου και από τον Επίτροπο. Αυτή ήταν έκθεση του Κοινοβουλίου που πήρε άλλη κατεύθυνση. Δεν καταφέραμε να, να έχουμε μια σχέση που θα μας συντόνιζε καλύτερα με την Επιτροπή. Κάτι που συμβαίνει κανονικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερο συντονισμό ε, είχαμε με το Συμβούλιο, το αντίθετο από ό,τι αναμενόταν. Διότι έπρεπε να επαρσιστούμε τι θέσει μα από τον Επίτροπο, με τον οποίο δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε. Το λόγιο, επειδή είμαστε κυκλισμένοι των θυρών. Ο συντονισμό εξαρτάται βέβαια και από τι προσεγγίσει. Αυτό επηρέασε κάπω και ότι κανένα από εμά δεν γνώριζε την όλη κατάσταση. Μαθαίναμε το πώ λειτουργεί στην απόφαση ενώ δουλεύαμε. Ε, και είχαμε την, αποκτήσαμε αίσθηση των δυνάμεών μας. Όχι αμέσως όμως. Σιγά σιγά καταλαβαίναμε ποια ήταν. Σήμερα μια μεταρρύθμιση της ΚΑΠ σίγουρα θα έπαιζε διαφορετικό ρόλο στο Κοινοβούλιο χάρη στην πρώτερη εμπειρία. Μάθαμε δηλαδή. Καταλάβαμε πώς να εκμεταλλευτούμε πλήρως τον ρόλο μας. Αυτά τα δύο στοιχεία ήθελα να τα υπογραμμίσω. Με άλλο επίτροπο που θα εκμεταλλευόταν των εισαγωγικών, που θα έπαιζε περισσότερο το χαρτί του Κοινοβουλίου σε κάποια μεγάλα ζητήματα που δεν αφορούσε συμφέροντα ε, κρατικά, αλλά συμφέροντα της Ευρώπης, ίσως διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζος Λάιον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ στη συνεδριασή της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και είχατε ευκαιρία εδώ μερικούς παλιούς φίλους. Θα προσπαθήσω να είμαι λιγάκι σύντομος. Για τις παρατηρήσεις του Ντεκάστρο, εγώ θα συμφωνούσα ότι η Ιρλανδική ε, Προεδρία ακολούθησε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε επίπεδο προσωπικών επαφών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι ότου φτάναμε στους επίσημους τριγωνικούς διαλόγους, η εντύπωση στο παρελθόν ήταν ότι η Κομισιόν δεν είχε καμία και το γραφείο του Αρμόδιου Επιτρόπου δεν είχε καθόλου επαφή με τους ε, βουλευτές. οι συζητήσεις όπου προσπαθούσαν να καταλάβουμε τι θέλανε, που ήταν οι κόκκινες γραμμές τους για να έχουμε μια καλύτερη ε, επαφή με την Κομισιόν. Ε, δεν ίσχυε στο παρελθόν, ενώ από την πλευρά της Ιρλανδικής Προεδρίας, από τη στιγμή που ο Σάμ Κόμετρη πήρε την ξεκίνησε στην Ελλαδική Προεδρία, υπήρχε μια απόλυτη σαφήνεια με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ξέραμε πολύ καλά ποιοι ήταν οι στόχοι, τι θέλαν να επιτύχουν οι βουλευτές από τη μία πλευρά και το Συμβούλιο από την άλλη μεριά και ο Σάιμον ο ίδιος έδειξε ένα προσωπικό ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα θέματα και προσπάθησε να έρθει σε επαφή με όλους. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον. Ένα από τα διδάγματα τα οποία πρέπει να αντλήσουμε ω Κοινοβούλιο είναι ότι όλο το θέμα των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών και της συναπόφασης <clears throat> ήταν θέματα τα οποία πολλές φορές είχαμε προσκρούσει σε τριγωνικούς διαλόγους που μας λέγανε ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση αυτά τα θέματα. Αυτό ήταν μια πραγματικά παράλογη θέση. Το συζητήσαμε στην ε, στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που θεωρήσαμε ότι υπάρχει κίνηση η διαδικασία των δημοσιονομικών προοπτικών να αποστέλει στο Κοινοβούλιο από τη δυνατότητα να συμβάλλει αποτελεσματικά σε ένα μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων. Για, τη, για τα θέματα αυτά λοιπόν του, των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο εναπέκειτο στους συζητητές των επιτροπών. Πρέπει λοιπόν την επόμενη φορά και αυτό δεν οδήγησε σε συγκροτημένη αντιμετώπιση. Πρέπει την επόμενη φορά λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί για τη διαδικασία που θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές γιατί αυτό αφαιρεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιαδήποτε δυνατότητα διαπραγμάτευση. Αν μα λέτε ότι δεν μπορείτε εσεί να αλλάξετε αυτό το οποίο έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό είναι απώλεια εξουσιών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάποια τελευταία σχόλια. Η έκθεση αυτή αναφορερόταν στην επιρροή των γεωργών στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι η έκθεση έχει την άποψη ότι οι προτάσεις της Κομισιόν ήταν οι ριζοσπαστικές προτάσεις μεταρρύθμισης και το Κοινοβούλιο τις αποδυνάμωνε. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή σωστό σημείο εκκίνησης. οι προτάσεις της Κομισιόν για μένα ήταν ιδιαίτερα άτολμες τις περισσότερες φορές για τα θέματα παραγωγής χάρη της κλιματικής αλλαγής. Πολλοί από εμά ζητήσαμε περισσότερη ευκαμψία για να μπορέσουν τα κρατημέλη να προχωρήσουν περισσότερο στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που είχε να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά τελικά καταλήξαμε με μια ενιαία λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα μέτρα τα οποία, στα οποία κατέληξε η μεταρρύθμιση δεν ήταν πάντα τα καλύτερα. Εγώ λοιπόν θα διαφυσβητούσα την ιδέα αυτή ότι η Κομισιόν είναι ο χρυσούς κανόν και η δική της πρόταση ήταν πιο φιλόδοξη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς την αλλίωνε. Αυτά λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Μα με ρωτήσατε και αυτό το ερώτημα για το ποσοστό επιτυχίας στην, ε, στον κανονισμό EFRD e σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές. Για μένα ήταν πιο εύκολο να βρούμε σε αυτό το θέμα μεγαλύτερη ευκαμψία γιατί δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, ενώ οι άμεσες πληρωμές ήταν ένα ιδιαίτερα πολιτικό, πολιτικοποιημένο θέμα και ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια κοινή συμβιβαστική λύση. Δεν υπήρχε πραγματικό περιθώριο έλιγμου και όλα αυτά είχαν κυρίως ε, σαν κέντρο την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών. Αυτά ήθελα να πω. Κύριος Κάπουλα Σάντους τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε, η οποία μου έδωσε μεγάλη χαρά και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να ξαναδώ παλιούς γνώριμους και που φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της έκθεσης για τη θαυμάσια αυτή η έκθεση που μας παρουσίασε. Τα τελευταία χρόνια η μονάδα Β μας έχει δώσει πολύ καλά έγγραφα εργασίας και από όλα αυτά αυτή την έκθεση θα τη διαβάσω με μεγαλύτερη προσοχή γιατί νομίζω ότι η τελική μου γνώμη για αυτή την εργασία είναι πάρα πολύ θετική. Συμφωνώ με τα περισσότερα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και θα σταθώ σε αυτές τις εξαιρέσεις. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Για εγώ ως συμμετέχον σε αυτή τη διαδικασία θέλω να σταθώ στην ε, άποψη ότι το Κοινοβούλιο ξεκινά από μια θέση εκκίνησης η οποία είναι μειονεκτική. Για δύο λόγους. Καταρχήν η θεσμική θέση των, συν, των ε, εισηγητών. Εγώ ως εισηγητής στο παρελθόν χρειάστηκε να συζητήσω με, τους ε, Ευρωπαίους, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Γεωργίας. <clears throat> και στη συνέχεια εγώ έπρεπε να παίζω τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συζητώ με τους εμπειρογνώμονες σε τεχνικό επίπεδο των άλλων θεσμικών οργάνων. Δηλαδή να συνδυάσω τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Θέλω να τονίσω και κάποιο άλλο σημείο που παραβλέπει αυτή η έκθεση. Σίγουρα ο, κύριος Σάιμον Κόβενι ήταν ένας από τους ήρωες της διαδικασίας της ε, μεταρρύθμισης, αλλά για μένα ο κύριος ήρωας ήταν η γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας που έπρεπε να αντιμετωπίσει τους υπερμηχανισμούς των, ε, της, του, της Προεδρίας και της Επιτροπής. Εγώ ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο ήταν τότε στην αντιπολίτευση της χώρας μου, δεν μπόρεσα να έχω την υποστήριξη από το Εθνικό Υπουργείο Γεωργίας που θα έδινε το ίδιο Υπουργείο σε ένα βουλευτή της κυβέρνησης σε έναν ευρωβουλευτή που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Και φυσικά δεν υπήρχε κανένα συμφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης της χώρας μου να υποστηριχθεί η δική μου εργασία και να παρουσιαστεί ως κάτι το θετικό γιατί αυτό θα ακύρωνε την επιτυχία που ήθελε να προσποριστεί η κυβέρνηση της χώρας μου. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να εγγραφεί στα συμπεράσματα αυτής της ε, έκθεσης είναι η ανάγκη να ξαναδούμε το θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου θα πρέπει οι εισηγητές του Κοινοβουλίου να βρίσκονται σε ίσο επίπεδο με τους ε, υπουργού και τους επιτρόπους και σε επίπεδο τεχνικών διαπραγματεύσεων να βρίσκεται κάποιος γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δεν έχουν την τεχνική ικανότητα οι, οι Εγώ εντάξει δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου αλλά έχω σταθεί ε, τεχνοκράτη στο Υπουργείο Γεωργίας της χώρας μου. Έχω μια προσωπική εμπειρία που μου επέτρεψε με κάποια δυσκολία να διεξαγάγω τη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο με τους γενικούς διευθυντές της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνεται με οποιοδήποτε βουλευτή. Αυτό είναι απόλυτα άδικο. Ένας οποιοδήποτε βουλευτής δεν μπορεί να περιμένει να είναι οι στα θέματα της γεωργίας για να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο και τις Κομισιόν που διαθέτουν τις πιο ισχυρές γραφειοκρατίες για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω και πάλι και μπορώ να το πω τώρα με μεγάλη ε, χαρά ότι για μένα αυτοί που ήταν οι πραγματικοί ήρωες της διαδικασίας ήταν οι συνεργάτες των βουλευτών και το πολύ περιορισμένο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σε συνθήκες άκρας ανισότητας μπόρεσε να ανταγωνιστεί την Κομισιόν και το Συμβούλιο με αποτέλεσμα για το οποίο δεν μπορούμε να ντρεπόμαστε. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε όπως είναι φανερό. Το Κοινοβούλιο μπόρεσε να περάσει πολλές από τις απόψεις του και αυτό φαίνεται και στα συμπεράσματά σας απόλυτα. Δύο ακόμα πράγματα θέλω να αναφέρω που διαφωνώ με την έκθεση. Λέει η έκθεση ότι η διαδικασία αυτή τελείωσε τον Ιούνιο. Όχι, το φθινόπωρο τελείωσε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέβαλε ότι αντίθετα με όλα αυτά τα οποία είπαν τα μέσα ενημέρωσης και η προπαγάνδα της Ιρλανδικής κυβέρνησης και θέλω να συγχαρώ την Μέρη Μαγκίνες για την ικανότητα της κυβέρνησής της στην επικοινωνία. Όλοι λέγανε ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν τότε τον Ιούνιο, αλλά οι αποφάσεις ελήφθησαν αργότερα. Μας υποχρέωσε το Συμβούλιο, όπως ε, ελέγχθη, να ακολουθήσουμε ορισμένες κατευθύνσεις, γιατί για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ουσιαστικά πήρε αποφάσεις σε επίπεδο θεματογεωργίας, ουσιαστικά παρακάμπτοντας τους δικούς του υπουργούς. Μας είπε ο Υπουργός της ε, Ιρλανδίας, της Γεωργίας, ότι τα θέματα αυτά του κάπινγκ και της μεταρρύθμισης δεν μπορούν να συζητηθούν πλήρως γιατί είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είχε ήδη σε συζήτηση τα θέματα αυτά. Υπήρξε λοιπόν μια σαφής ανισότητα όπλων στη διαπραγμάτευση αυτή που έκανε ακόμα πιο δύσκολο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν το μέλλον. Έχω κλείσει λοιπόν ένα ακόμα θέμα ε, με το οποίο δεν συμφωνώ απόλυτα είναι το ότι λέγεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μείωσε το greening. Όχι δεν είναι αλήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αδύνατο να γίνει μια πρόταση η οποία ήταν μη ρεαλιστική. Ακύρωσε τις προτάσεις της Κομισιόν που ήταν αντιρεαλιστικές. Αν τώρα έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μία εφαρμογή του greening είναι γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει η Κομισιόν η οποία θα είχε αυτοακυρωθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους. Και ευχαριστώ και την Πορτογαλική καμπίνα που έχω πολύ καιρό να τη δω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια γενική ανάλυση που δεν μπορούσε ε, να εξαχθεί από την έκθεση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ο ανθρώπινος παράγων αναφέραμε το όνομα Υπουργού Ιρλανδού. Ε, βεβαίως αυτή η Προεδρία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Έφτασε στην Προεδρία ε, με την βούληση να επιτύχει και όλες οι υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν γι' αυτό. Ο χρόνος στον οποίο βρεθήκαμε, λοιπόν, η χρονική στιγμή ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είχαμε δει με προηγούμενη Προεδρία ότι είναι αδύνατο να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία. δεν ήταν δυνατόν με την προηγούμενη Προεδρία να γίνει μεταρρύθμιση. Μετά έχουμε τυχαία γεγονότα. Κάτι τυχαίο. Ήμασταν από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι οι τρεις εισηγητές και ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας μπόρεσαν να συνεννοηθούν. Ε, δεν κατόρθωσε τίποτε να μας διαιρέσει όταν ήμασταν σε δύσκολες στιγμές και σε στρατηγικές στιγμές. Ίσως να ήμασταν τυχαία ίσως και οι τέσσερις από χώρε της Νότιας Ευρώπης. Είχαμε και οι τέσσερις ίσως την ίδια θεώρηση της Γεωργίας, το βλέπουμε στην εισήγηση. Ε, η διαίρεση έγινε, η διαφορά έγινε ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Νομίζω ότι στο μέλλον σε εισηγήσεις τόσο σημαντικές δεν θα πρέπει απλώς να ορίζονται εισηγητές, αλλά επίσης να υπάρχει μια ομάδα εισηγητών ε, η οποία να μπορεί να συνεργάζεται, ε, να είναι ενωμένη απέναντι στο Συμβούλιο και στην Επίτροπη. Αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη. Και μετά και αυτό λέχθηκε από τον συνάδελφο Βίσκ. Εγώ θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, στην εργασία των ατόμων που μας βοήθησαν. Η βοηθή μας πρώτα απ' όλα. Ο βοηθός μου κάποια στιγμή νόμιζα ότι επρόκειτο να εκραγεί οι υπηρεσίες της γραμματείας ε, που, στις οποίες ασκήσαμε πάρα πολύ πίεση και οι άλλοι διαπραγματευτές ε, θα χρησιμοποιούσαν το παραμικρό μας λαθάκι αν μπορούσαν για να κερδίσουν στο παιχνίδι ρόλων που είχαμε. Αλλά Είπα και στην Επιτροπή Γεωργίας ότι για σημαντικές εκθέσεις όπως αυτήν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξοπλίζεται για να μπορεί να στηρίξει διοικητικά την ομάδα τη διαπραγμάτευσης. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός νομικού κλπ. Πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη ομάδα που να συνοδεύει τον εισηγητή και να κάνει την εργασία μαζί μας. Για το φάκελο τώρα της κοινή οργάνωσης αγοράς. Σήμερα, 18 μήνες μετά και σε σχέση με όσα βλέπουμε να φτάνουν στην Επιτροπή Γεωργίας, κατανοώ ορισμένα πράγματα. Η έκθεση αυτή ήταν μια συναρμολόγηση, ένα συνονθήλευμα ε, κειμένων που δεν ήταν έτοιμα στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και που η Κομισιόν δεν είχε πρόθεση να διαπραγματευτεί στα πλαίσια της ΚΑΠ. Ενώ διαπραγματευτήκαμε πριν από 1,5 χρόνο, βλέπουμε σήμερα μια έκθεση για το, τα γαλακτοκομικά, την προοπτική μιας έκθεσης για την κοινή οργάνωση αγοράς για τα φρούτα. Τι να πούμε για τον Ίνο, όπου χρειάστηκε να αγωνιστούμε θα πρέπει επίσης στο μέλλον η Κομισιό να έρχεται να διαπραγματευτεί με έτοιμους φακέλους γιατί χρειάστηκε να γίνει μια εργασία γραφής και νέας γραφής αναδιατύπωση με ε, κείμενα τα οποία δεν είχαν συνεκτικότητα μεταξύ τους, διότι ήταν ένα συνονθήλευμα κειμένων που δεν είχαν σύνδεση μεταξύ τους. Προσωπικά ήταν για μένα καλή εμπειρία, καλή ανάμνηση και κακή ίσως από την πίεση, αλλά είχα την εμπιστοσύνη σας για αυτή την έκθεση. Ναι. Τρία άτομα θα ήθελα να, λάβουν τον λόγο, η κυρία Ιουσέ, ο κύριος Φερό η ε, κυρία. και η κυρία Μαγκίνας. Δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νέα βουλευτής, Επομένω δεν ξέρω πολύ καλά αυτή τη διαδικασία, δεν έχω ενταχθεί σε αυτήν. Την έχω παρακολουθήσει όμως από έξω κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν να κάνουν όχι με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων αλλά με τον τι ακριβώς και πώς έτυχε διαπραγματεύσεων. Δεν βλέπω τώρα όπως ο προλαλής σας ίσως το κοινοβούλιο σαν ένα μονολυθικό σώμα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς θα έπρεπε να είχε γίνει η μεταρρύθμιση στην αγροτική πολιτική. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες ήταν οι πολιτικές οικογένειες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία. Υπήρξαν κάποιες ομάδες οι οποίες μπόρεσαν να περάσουν με επιτυχία τις ε, θέσεις τους ή υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν το κατάφεραν καθόλου. Φυσικά είμαστε κομμάτι μιας μεγάλης ομάδας, αλλά ήταν και ομάδες οι οποίες είχαν συγκεκριμένες απόψεις για τα θέματα αυτά και θέλησαν να τις περάσουν. Με ενδιαφέρει επίση το θέμα της, των εισηγητών. Είπατε, αν η προσωπικότητα του εισηγητή παίζει μεγάλο ρόλο για την ε, επιρροή που μπορεί να ασκούσει να ασκήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φυσικά τότε είναι πάρα πολύ σημαντική η επιλογή των εισηγητών και δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη και δεν πρέπει να αφήνεται μονάχα σε επίπεδο προσωπικών συμφερόντων, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε με πολύ μεγάλη προσοχή ποιος παίρνει την κάθε έκθεση και επομένως είναι μια προϋπόθεση για ένα καλό αποτέλεσμα η ε, επιλογή των εισηγητών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, να γνωρίσω από εσά τι ρόλο παίζει ο εισηγητή και πώς έχουν, τι αποτελέσματα έφεραν τα συγκεκριμένα κόμματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το σεμινάριο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας επιτρέπει ε, να δούμε μετά από έξι μήνες, να κάνουμε μια ανασκόπηση ε, μετά από έξι μήνες θητείας του νέου κοινοβουλίου. Το σεμινάριο αυτό θα μπορούσε να γίνει στα Ανάντι Δηλαδή νομίζω ότι οι ομιλητές σήμερα το πρωί είδαν ότι θα πρέπει στα ανάντι να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην Κομισιό και αυτό φτάνει ίσως ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά αυτό που γίνεται τώρα και θα πρέπει βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξαναναλάβει τον ρόλο εξουσίας που έχει για να ετοιμάσει καλύτερα ε, την επόμενη ΚΑΠ είναι ένα θέμα κυριαρχίας, μια πράξη κυριαρχίας. Σήμερα πρέπει να ξαναδώσουμε το λόγο στο λαό και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να μπορεί να προτείνει τα μέσα, τα εργαλεία για μια καλύτερη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη. Σχετικές με τις τροπολογίες, εγώ είμαι μη εντεταγμένος, μη εγγεγραμμένος βουλευτής και δεν έχω πρόσβαση στις εκθέσεις. Έκανα δύο αιτήσει που και μου αρνήθηκαν την πρόσβαση και νομίζω ότι ε, το καπηλεύονται ορισμένοι το κοινοβούλιο. Θα, αν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε ευροσκεπτικιστές βουλευτές, θα πρέπει να συνεχίσετε να μας αποκλείετε για τις τροπολογίες και για τις εκθέσεις. Είναι δύσκολο λοιπόν να επιζήσει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Σχετικά με την ουσία, ο ε, κανονισμός σήμερα είναι η οδός της νέας ποιος είναι ο στόχος να ρυθμίσει για να ρυθμίσει, για να ρυθμίζει. Θα πρέπει να αποφύγουμε ε, μεγάλες κρίσεις να μην ε, καταστρέφουν τον μηχανισμό παραγωγής και οι μηχανισμοί για την επεξεργασία της νέας ΚΑΠ 2014-2020 βασίζεται στην διάρθρωση των αγορών απέναντι στις αγορές, στους βιομήχανους και στην ε, διανομή, στην εμπορία. Οι μηχανισμοί αυτοί ποικίλουν κυρίως όταν είναι σημαντικοί ακόμα και όταν οι κίνδυνοι είναι μικροί γιατί πρέπει να εξαρθόμαστε από τις οργανώσεις παραγωγών που δεν μπορούν ε, να αντιμετωπίσουν διεθνείς ε, συνομιλητές, όλο και πιο σημαντικούς. Δεν έχουν κανένα μέσο να καταπολεμήσουν το κοινωνικό dumping και τις πτωτικές τιμές σε περίπτωση κρίση. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, διότι ε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την παρατεταμένη πτώση των τιμών. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι εμείς οι αιρετοί καθόμαστε και ακούμε τους συμβούλους να μιλάνε για, προ, για πρασίνισμα, για αναλογικότητα. Αλλά οι αγρότες έχουν δυσκολίες και το Δεκέμβριο 2014 θα έχουν ζημίες και όσους μακριά από αυτό το ημικύκλιο ε, καταραίουν λόγω αυτής της ΚΑΠ και λέω κύριε Πρόεδρε ότι καθισμένοι εδώ, ακόμα και αν οι μελέτες είναι, είναι ε, σημαντικές, είμαστε ε, σαν τους Βυζαντινούς που συζητούσαν για το φύλλο των αγγέλων όταν έπεφταν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Αντιπρόεδρε Μαγκίνες, έχετε το λόγο. Δύσκολο από πού να ξεκινήσω. Έχω δύο λεπτά στη διάθεσή μου. Πρώτα απ' όλα κατά κάποια έννοια θα ήταν ευκολότερο να είμαστε εκτός διαδικασίες. Ε, άλλοι συνάδελφοι εξέφρασαν απόψεις. Να συγχαρούμε αυτούς που ενεπλάκησαν εμάς και τους ηγητές που εργαστήκαμε πολύ σκληρά και καταλήξαμε σε αποτέλεσμα. Ε, πανεπιστημιακός και πολιτικός κόσμος είναι διαφορετικός, αλλά άδει και νερό. Και να σας πω ότι η πρακτική εφαρμογή των πολιτικών για τις μεταρρυθμίσεις ήταν κάτι πρωτόγνωρο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο διαπραγματεύσει σε κάθε επίπεδο ε, έκανε πολλή δουλειά η γραμματεία της Επιτροπής ε, Γεωργίας και η βοηθή μας ε, πολύτιμη, πολύ πολύτιμη εργασία. Δεν μπορούμε να συγχαρούμε αρκετά για ό,τι κάνανε. Εγώ σε τι ενοχλήθηκα όσον αφορά τη μετάσταση της ΚΑΠ. Στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνομιλήσε αρκετά καλά με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις διαβουλεύσεις είχαν έτοιμα τα έγγραφά τους, κατά την απόψή μου, ε, ήξεραν τι έρχεται και δεν συζήτησαν με τους πολιτικούς. Ε, δεν μας είπαν τι είχαν υπόψη τους, δεν μας ενημέρωσαν έγκαιρα και σπαταλήσαμε πάρα πολύ χρόνο και προσπάθειες. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής μας, ο οποίος αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν κάκιστες. Ε, και αυτό έπνιξε τις άτυπες διαπραγματεύσεις και δεν μπορείς να τις αποτιμήσεις, ούτε μπορείς να αναφέρεις εκθέσεις αυτές, αλλά είναι πραγματικά σημαντικότατες. Το ζήτημα για τη μεταρρύθμιση της κάποιο ήταν. Πάντα όλα ήταν μπερδεμένα. Θέλαμε να δώσουμε δημόσια χρήματα ή δημόσια αγαθά και ο ορισμός των δημοσίων αγαθών ε, δεν είναι κάτι προσμετρήσιμο και ξεκάθαρο και συμφωνώ με τον εισηγητή. Την αποδυνάμωση ε, της προσπάθειας. Είναι το, υποκειμενικό. Αν λέγαμε αλλαγή, εντάξει, να πούμε αποδυνάμωση, είναι υποκειμενικό. Και ακολουθεί η πολιτική γραμμή συγκεκριμένη που δεν δέχομαι. Στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με τη δυσχέρεια εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που διαπραγματευτήκαμε. Είναι πολύ δυσκολή αυτή η πολιτική θέση στην οποία βρισκόμαστε είναι το θέμα το σημαντικό των κατεξοδότησης πράξεων και ακόμα δεν είδαμε πώς θα εξελιχθεί συνοπτικά. Θαύμα αυτό που πετύχαμε. Ήταν η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο είναι πλάκι και τα λόμπι των γεωργών δεν συνομίλησαν καλά με το κοινοβούλιο, κάναν τα κολπάκια τους με την Κομισιόν. Δεν έδειξαν σεβασμό προς το κοινοβούλιο. Ναι, πολλά μαθήματα μπορούμε να μάθουμε. Μου ξύπνησαν εφιάλτες για μένα και όχι όνειρα, γιατί ήταν εφιαλτική κατάσταση για μας που εργαζόμασταν. Δεν μπορούμε να προβούμε σε τελική αξιολόγηση μέχρι ότου δούμε την εφαρμογή. Αλλά βλέπω ότι σηκώνει το σφυράκι σας, Πρόεδρε, οπότε θα σταματήσω. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σίσλινγκ. Πρέπει να σκεφτούμε, λέει ο κύριος Χόισλινγκ, να δούμε πόσο εκπληκτικό είναι το ότι καταλήγουμε τελικά σε μια συμβιβαστική λύση. Βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ξεκίνησε από την απόλυτη απόρριψη της πρότασης του Κομισιόν και σιγά σιγά καταλήξαμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων η οποία οδήγησε σε κάποια συμφωνία στο τέλος. Αυτό δεν τα κάτι που μπορούσε το να προστοκά εξ αρχής. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του ρόλου του εισηγητή. Είναι ένας πράγματι προεξάρχων ρόλος και φυσικά η ικανότητα του εισηγητή να πείθει τις άλλες πολιτικές ομάδες δεν φτάνει να πει ότι αυτή είναι η θέση μας και τελείωσε. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία. Όλα θα μπορούσαν να είναι κάπως καλύτερα φυσικά, αλλά γενικά νομίζω ότι υπήρξε ένας πολύ καλός δρόμος που ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελικά μπόρεσε να καταλήξει σε μια ενωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά έρχομαι πάλι στο θέμα του ρόλου του Κοινοβουλίου ως σύνολο. Ελέγχθη ότι εμείς είμαστε εκπρόσωποι των γεωργών και είμαστε εκπρόσωποι των αγροτικών συμφερόντων σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η πραγματικότητα. Εμείς ως Αγροτική Επιτροπή δεν είμαστε μονάχα οι εκπρόσωποι στενών συμφερόντων των γεωργών. Εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη το γενικότερο πλαίσιο και όχι να θεωρούμαστε ότι είμαστε μονάχα εκπρόσωποι των γεωργών. Το θέμα είναι λοιπόν <clears throat> και πώς γίνονται οι συμβιβαστικές λύσεις. Με τον Επίτροπο Τσόλος στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι απόψεις. Και παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν υπήρξε συμφωνία υπήρξε συνεννόηση μεταξύ μας, οι ίδιοι οι κοινοβουλευτικοί οι οποίοι κατάφεραν να έχουν αυτές τις συμβαστικές λύσεις, μετά βγαίνανε πολλές φορές και λέγανε ότι εγώ ήμουν εναντίον από την αρχή και ήταν κακή η μεταρρύθμιση κτλ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα, η μεταρρύθμιση σε αυτή την περίπτωση, να την χάνει και αποδοχής. Όποιος λοιπόν συμβάλλει σε μια συμβαστική λύση έχει την ευθύνη να την να πείσει και τους άλλους για τη σημασία αυτής της λύσης. Θα πρέπει λοιπόν να φέρουμε το βάρος των αποφάσεών μας και να όχι να λέμε στη συνέχεια ότι αυτά δεν είναι σωστά και θα έπρεπε να τα είχαμε απορρίψει όλα. Αυτό μπορεί να κερδίζει υποστήριξη σε πολιτικό επίπεδο και να έχει καλούς πηχαίους τίτλους σε εφημερίδες, αλλά δεν Μα πηγαίνει πουθενά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε και μια σαφέστερη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η Κομισιό θα μα δίνει πάντα κάτι το οποίο μα ικανοποιεί απόλυτα. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ε, μεταρρύθμιση με τον δικό μα ενεργό τρόπο, λαμβάνοντα πλήρω μέλο σε όλε τι συζητήσει και διαπραγματεύσει. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριος Νταντέ. Δύο λεπτά. Εδώ κάνουμε απολογισμό της μεθόδου και κάνουμε προτάσεις. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης δεν ολοκληρώθηκε, και οι της συμπράξεις δεν έχουν εκδοθεί όλες. Ε, εγώ κάνω την πρόταση, Προέδρε, που θα πρέπει να συνδέεται, ε, να συζητηθεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να παραμείνει για να παρακολουθήσει την εφαρμογή των κατοξιδότητες συμπράξεων. Βλέπουμε και με τα δικαιώματα τα φυτεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Χρειάζεται συνομιλητές οι οποίοι επίσημα να καθορίζονται. Η διαπραγματευτική ομάδα των εκθέσεων θα πρέπει να φτάσει μέχρι τέρμα, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για τις κατεξουσοδότης πράξεις. Ο Πρόεδρος πέρασαν τα δύο λεπτά. Και τώρα είναι η δική μου σειρά να μιλήσω και εγώ για δύο λεπτά γιατί και εγώ είναι πλάκιν στην όλη προσπάθεια. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι έλειπε το σφαιρικό όραμα. Ε, είχαμε ένα συνονθήλευμα ιδεών και ε, ανεπαρκής εμβάθυνσης από πλευράς Κοινοβουλίου επίσης υπήρξε. Ήταν η πρώτη φορά παρόλα αυτά παρά την ε, σοφία και την επιδεξιότητα των Ευρωβουλευτών δεν ήμασταν η καλύτερη διαπραγματευτική ομάδα που μπορούσε να υπάρξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριεφέρθη όπως συνήθως. Ο Επίτροπος άκουσε, μας άκουγε, συμφωνούσε και μετά έκανε τα δικά του. Ε, νομίζω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πολλά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Χθες κατέστησα φες ότι ο Επίτροπος πραγματικά έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου από τους δημόσιους υπαλλήλους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε την ΚΑΠ και μας είπαν ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το πρασίνισμα, διότι χωρίς πρασίνισμα δεν θα υπήρχε ΚΑΠ. Αυτό όμως δεν αληθεύει. Βέβαια έχουμε την κρίση, έχουμε δημοσιονομικές πιέσεις, 40 δισεκατομμύρια λιγότερα για την ΚΑΠ, Και μετά είναι και όλη η συζήτηση για την κοινοτική μέθοδο έναντι διακυβερνητικής μεθόδου. Δεν μπορούμε τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες για όλα αυτά. Στην όλη αυτή λοιπόν κατάσταση που επικρατεί, εμείς κάναμε διάφορες παραχωρήσεις. Θέλαμε να υπερασπιστούμε την κοινή αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι θα θυμόσαστε όλες τις, την πάλι την διαπάλη μεταξύ πολιτικών ομάδων για την ανάθεση των εκθέσεων. Τελικά όμως συνεργαστήκαμε καλά και όλοι έλαβαν υπόψη τις ιδέες άλλων, οι μεν τις ιδέες των άλλων. Η Αντιπρόεδρος Μαγκίνες φρόντισε τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών έτεινε νεβίκον ους προς τις ανάγκες αυτές. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την ε, ενσωμάτωση διαφόρων τροπολογιών στο κείμενο. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε τα μαθήματά μας, μας το είπε άλλωστε ο κύριος Νταντέ. Ε, τα υπόλοιπα στοιχεία των μεταρρυθμίσεων καλύπτονται από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Έχουν αυτή τη μορφή και θα πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό πριν γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση. Για να δούμε, μου έδωσαν κάποιο σημείωμα να δώσω το λόγο τώρα στον καθηγητή Σουίνεν. Αν θέλετε καθηγητά να απαντήσετε στα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον Ατήλα, διότι υπήρξε ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι και εύκολο να απαντηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τις ομάδες, το ΕΛΚ ήταν οι πιο επιτυχής, μετά σοσιαλιστές και οι πράσινοι, μετά οι μία γεγραμμένοι είχαν τις λιγότερες επιτυχίες. Αυτά όσον αφορά τα ποσοστά των επιτυχιών των ε, πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα άλλα σχόλια. Δεν νομίζω είναι ορισμένα πράγματα που ήταν πάρα πολλά χρήσιμα, χρήσιμες ε, δηλώσεις και όχι απαραίτητο ε, σχόλια για την έκθεση, ήταν μάλλον για την όλη διαδικασία. Εγώ θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που επανήλθαν, επαναλήφθηκαν από πολλά άτομα ίσως ε, ως προς τη διατύπωση ορισμένων θεμάτων, την αντίληψη ε, της, ε, του περιορισμού του πρασινίσματος, της αποτυχίας του πρασινίσματος. Δύο φορές είπα στην μελέτη ότι η αντίληψη του status quo και της μεταρρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό, αν παραδείγματο χάρη η Κομισιό μας πει, όχι, με συγχωρείτε, αν ένα άτομο πει ότι θέλουμε να επανεισαγάγουμε μια κάποια διασύνδεση, να έχουμε ε, μια κατάσταση που δεν θα υπάρχουν, δεν υπάρχει αποσύνδεση και decoupling. Αυτό είναι status quo ή είναι μεταρρύθμιση. Από αυτήν ε, την ε, άποψη, αν νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσετε έτσι, αυτό είναι status quo και η νεοφιλελεύθερη για την νεοφιλελεύθερη είναι το status quo αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όσοι νομίζουν ότι πρέπει να υπάρχει υπάρχει επανασύνδεση για να αντιμετωπίσουμε την πτώση των τιμών, τότε είναι μεταρρύθμιση. Προσπαθούμε να απαλλαγούμε από αυτές τις αντιλήψεις και νομίζω ότι για το greening προσπάθησα να κάνω το ίδιο. Θα ελέγξω και πάλι ε, πως αυτή η αντίληψη του watering down ε, είναι σωστή ή όχι. Παραμετός χάρη Νομίζω και αυτό λέχθηκε και στις συνεντεύξεις ότι δεν θέλαμε να μειώσουμε το πρασίνισμα, θέλουμε να ακολουθήσουμε τρόπους διαφορετικούς, πιο βιώσιμους, πιο πρακτικούς. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν ακούστηκε η παρέμβαση. Έχουμε στο κείμενο ε, το, το πρασίνισμα είναι κάτι το σφαιρικό, είναι κάτι το γενικό και λέμε ότι για ορισμένα πράγματα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να προχωρήσει περισσότερο από την πρόταση της Κομισιόν. σω μερικά πράγματα ε, χάθηκαν ίσως ε, καθοδόν. Στο ίδιο ισχύει για την αντίληψη του αγροτικού συμφέροντος, agricultural interest. Νομίζω ότι στην ίδια την έκθεση ε, τεκμηριώνουμε τι εννοούμε με αυτό, με την έννοια ότι λέμε από τη μία πλευρά ότι υπάρχει η αντίληψη αυτή, αλλά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να σταθμίσουμε, να μετρήσουμε. Νομίζω ότι το βασικό σημείο εδώ δεν είναι αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει, είναι πώς άλλαξε με την συναπόφαση. Ε, η προσμονή, η προσδοκία ήταν ότι διαφορετικά άτομα θέλανε ε, να μπουν ε, στη μέση λόγω των διαφορετικών επιδράσεων και δεν το βρήκαμε αυτό τα άτομα με την ίδια βάση, το ίδιο background. Αυτό είναι το βασικό σημείο. Νομίζω το αναφέραμε αυτό σε σχέση με την Γεωργία. Είναι καλά προσδιορισμό το τελευταίο μου σημείο, διότι θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο για τα θέματα ε, προσωπικότητας. Αυτό είναι σημαντικό. Το ξέρετε αυτό. Το θέμα που μπορείτε να διαρωτηθείτε εάν ε, η ενδιάμεση αξιολόγηση θα μπορούσε να είναι εφικτή αν το αποτέλεσμα θα ήταν ε, διαφορετικό με άλλο αν ήταν ο Τσόλος ο Επίτροπος. Νομίζω ότι όλοι έχετε συγκεκριμένες απόψεις για το θέμα. Και ο ε, κύριε Ντεκάστρο, ναι, ε, θα έκανα μια άλλη έκθεση για την επίπτωση των άμεσων πληρωμών πάνω στη γη, στην αγορά και Θυμάμαι ότι στο Λουξεμβούργο κάποιος είπε, νομίζω κυρία Μαγκίνες, ότι όλοι θα έπρεπε να πάρουμε το λεωφορείο για το Λουξεμβούργο. Εκεί ε, σας αφήνω με αυτήν την σκέψη, διότι εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα για το θέμα αυτό. Ένα λεπτό κύριο Λάιον. το θέμα των συμφερόντων των γεωργών. Όταν λέτε πόσοι από τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας προέρχονται από το χώρο της Γεωργίας. Αν δείτε την Επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα βλέπατε εκεί πόσοι από αυτούς που είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουν ένα ε, μια τέτοια προέλευση. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό. η βασική ε, εντύπωση ήταν ότι η δική μας επιτροπή θα είναι προκατηλημένη και θα εκπροσωπεί μονάχα μία άποψη. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απόλυτα σωστό. Δεν είναι αξιόπιστη αυτή η αντιμετώπιση για το ρόλο της Επιτροπής μας. Θα κάνετε το ίδιο και με τις άλλες επιτροπές δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα, θεωρείτε, θεωρούσατε ότι και αυτές έχουν επεδεδημένα συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. εντάξει, ας μην πούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και προσβλέπουμε στην τελική ε, μορφή της έκθεσης αυτής και όπως είπε και ο κύριος Καπόλας Σάντος θα τη διαβάσουμε πολύ προσωπικά και θα πάρουμε τα απαραίτητα διδάγματα. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Καπούλας Σάντος. Απλώς θα ήθελα να πω το εξής. Το θέμα του τεχνικού προσωπικού της Επιτροπής Γεωργίας θα μπορούσε να ε, λυθεί χωρίς να υπάρχει πρόσληψη περαιτέρω προσωπικού αν για κάθε σημαντική έκθεση αποσπούνται από την Κομισιόν άτομα που έχουν την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Δηλαδή να ζητήσουμε από την Κομισιόν άτομα τα οποία θα λειτουργήσουν ως συνεργάτες του Κοινοβουλίου ακολουθώντας την ε, κατεύθυνση του Κοινοβουλίου. Αν είχαμε λοιπόν τεχνικό περι, προσωπικού σε όλες αυτές τις σημαντικές εκθέσεις, εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος και μόνος εισηγητής που θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο ισότητος με τις προεδρίες και με την ε, Κομισιόν. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ένας μονάχα εκπρόσωπος Συμβουλίου, ένας της Κομισιόν και πολλοί εισηγητές από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προ το παρόν αυτό δικαιολογείται επειδή δεν έχουμε το τεχνικό προσωπικό που να επιτρέψει σε ένα εισηγητή να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά τα θέματα. Αν έχουμε όμω την τεχνική ικανότητα θα ήταν καλό να έχουμε ένα ενιαίο εισηγητή και αυτό θα ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη που σα καθυστερώ περαιτέρω. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, και κάτι για μας να το σκεφτούμε και να το αναλύσουμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα να σκεφτόμαστε που αφορούν ε, το μελλοντικό μας ε, έργο. Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή τους. Αυτό που μάθαμε σήμερα ε, αξίζει τον κόπο να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ τους φιλοξενούμενους μας, τους καλεσμένους, τον κύριο Λάιν, τον κύριο Καπούλα Σάντος και όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.